we Να ξεκινήσουμε αν θέλετε, να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε βαρύ πρόγραμμα, φορτωμένο. Καταρχάς έχουμε ψηφοφορία με τον κύριο Σδρουγεύσκη για τις ε, τροπολογίες του προϋπολογισμού. Μετά έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό παιδείας και πολιτισμού του Λουξεμβούργου και θα συνεχίσουμε με την γνωμοδότηση επί των δημοσιονομικών. Ήθελα απλώς να πω εισαγωγικά ότι είχατε τα συμπεράσματα των ε, συντονιστών εχθές και θα ήθελα να τα εγκρίνουμε για να πάμε στο σημαντικό σημείο της πρώτης έκθεσης πρέπει να ψηφίσουμε και ευχαριστώ τη συνάδελφο ε, Σοϊντρόβα για την ε, πρόθεση της ε, επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Μαραγκάλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το προϋπολογισμό καθότι μόλις λάβαμε την έκθεση κομισιών για τα πιλωτικά. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο χρόνο να συναντηθούμε, να καταλήξουμε σε κάποιες θέσεις και να ψηφίσουμε στο τέλος. Χάνουμε εδώ το μικρόφωνο του ομιλητή. Sì, è vero, noi abbiamo ricevuto solo... Ναι, πράγματι εχθές το βράδυ αργά λάβαμε τις πληροφορίες αυτές, το οποίο είναι λίγο προβληματικό. Όμως εντός της ημέρας πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό να είναι σαφές για όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ας ε, τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες ομάδες, λοιπόν, παρακαλώ, και ο εισηγητής και θα δούμε τι θα προκύψει, θα λάβουμε μια απόφαση, αλλά επαναλαμβάνω, εντός της ημέρας πρέπει να ψηφίσουμε. Ο κύριος Μόργανο, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ένα τέταρτο για να δούμε αυτό που λέει ο συνάδελφος Μαραγκάλ, ένα τέταρτο 20 λεπτά τέλος πάντων, ώστε οι σκιώδεις μαζί με τον ε, εισηγητή να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Δηλαδή το να μην κάνουμε καμία επιλογή θα σήμαινε ε, να μην τοποθετηθούμε καθόλου σε επιτροπή. Βεβαίω. Εγώ θέλω να ακούσω και τι άλλε ομάδε, λέει η πρόεδρο. Μία δυνατότητα θα μπορούσε να είναι τώρα να ψηφίσουμε την έκθεση Σοϊντρόβα. Ναι, βεβαίω να ακούσουμε του προπολογισμού και να ακούσουμε και του υπουργού κτλ. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ακούσω του ηγητή και τι άλλε ομάδε. Κοιτάξτε πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν είναι 15 και 30 λεπτά να είναι. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά όπως είπε η πρόεδρος πρέπει να το κάνουμε σήμερα διότι διαφορετικά θα αποσταθεροποιήσουμε την όλη δουλειά της Επιτροπής. Penso che la, mm, difficile dire un quarto d'ora perché... Τώρα ένα τέταρτο είναι δύσκολο γιατί τώρα έχουμε Σοϊντρόβα, μετά καταφθάνει η Προεδρία του Λουξεμβούργου, πρέπει να είσαστε όλοι εδώ. Σας ζητώ επομένω, στις 12 το μεσημέρι να περάσουμε στην ψηφοφορία του προπολογισμού. Γιατί τα 15 λεπτά δεν ξέρω τώρα πώς θα, πώς θα γίνουν ακριβώς, γιατί στο μεταξύ θα πρέπει να ψηφίσουμε. Άρα δεν είναι 15 λεπτά. Ας πάμε στην ε, γνωμοδότηση. Σοϊντρόβα. Κάποιος λέει κάτι εκτός μικροφώνου. Δεν είναι τόσο ευγενικό, απαντάει η πρόεδρος. esattamente. Allora andiamo avanti, allora eh, Λοιπόν, θα κάνουμε αμέσως τώρα την γνωμοδότηση Σοϊντρόβα, Μόργανο, αλλά στη χειρότερη των περιπτώσεων στις 12 το μεσημέρι να, να έχουμε ολοκληρώσει το θέμα αυτό. Και κατανοώ το αίτημα γιατί η Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων πρέπει να τοποθετηθεί υπό το φως ε, των ε, περικοπών του Συμβουλίου. Άρα ψηφίζομαι ε, την γνωμοδότηση Σοϊντρόβα. είναι προφορική 3, μάλλον. Η τροπολογία 93 που έχει τροποποιηθεί από την 3 υπέρ, κατά, αποχές. 95 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. απορρίτεται 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 που έχει τροποποιηθεί από την προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Υπέρ, ε, η 106 με συγχωρείτε, υπέρ, κατά. Η συμβαστική 5 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100, όχι, συγγνώμη. Πάμε στην 113. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές Ελέγχουμε. Ελέγχουμε παρακαλώ. Okay. Uh, sorry. <laughs> I open the vote. I close the vote. Πέρασε ψηφοφορίας. Λέει τώρα η πρόεδρος. Όχι, όχι. Ακόμα ανοιχτή είναι. Ακόμα ανοιχτή είναι. Okay, That's, it does work. Yeah. This machine doesn't work. So can we... Μάλλον δεν δουλεύει το σύστημα. Ξανοίγουμε την ψηφοφορία. Okay, we reopen now the vote. τώρα την ψηφοφορία. Και πέρα στις ψηφοφορίες. Is rejected. Απορρίπτει. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτει. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχει ζητήσει το ΕΛΚΑ χωριστή ψήφο από τις 122 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται χωριστή ψήφος 141 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές για μένα εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος αλλά ας ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα Πέρα στις ψηφοφορίες. Μάλιστα. Απορρίπτεται λοιπόν. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 Χιούτσουκ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 155. Υπέρ. Όχι. Ναι, υπέρ. Κατά αποχές ε, πάλι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 156. Ταυτόσημη. Ταυτόσημη. 160. Όχι, όχι λέει πρόεδρος. Έχουμε γλωσσικό εδώ. 159. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 καταπίπτει. Πάμε 169 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 4, δηλαδή 173 τροποποιημένη από την προφορική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 174. Όχι. 170. 170. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 174. Υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ελέγχουμε για την 174. Παρακαλώ. I close the vote. ψηφοφορίας απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 πολύ σιγά πάμε λέει η πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 100, ναι εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημειώστε τώρα ότι η προφορική 5 επί 199 διαγράφει το very και προσθέτει το solely. Σημειώστε. Άρα επ' αυτού ψηφίζουμε χωριστή ψήφος για το, πρώτο το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 13 υπέρ. Όχι, όχι, χωριστή ψήφος ζητάει το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Εμπλ 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εμπλ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έμπλ 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται χωριστή ψήφο στο 210 που ζητάει το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία. Uh, sorry, I close the vote. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.13 λέει πάλι πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην MP1 κατά τμήματα, κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. MP2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. MP5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MP6 υπέρ κατά αποχές υπέρ εγκρίνεται, εγκρίνεται. MP8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. MP9 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 12, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 14, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 15, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 17, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 7 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τη λογική σκέψη Α7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Ετυλογική σκέψη Α8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ α υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλ d υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εμπλ ε κατά πίπτη. Περνάμε στην 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη D27. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 27. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά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 Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 1. MPI. I, λατινικό, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 42, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46. Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Σαράντα έξι. Όχι, όχι, λέει η πρόεδρος, ψηφίζουμε την ΕΜΠΛ ΚΑΠΑ. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56. Νέκοφ. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι, ποιος είναι κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 60. Πέρας. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63, 65, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη J, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλη L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη B υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη G υπέρ. Θέλετε να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος στην Έμπλη Β. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Έμπλη Β. Πέρας εγκρίνεται. MPG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Εβδομήντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. MPH. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εμπλη F υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη W υπέρ. Ε, τροπολογία 88. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 89. 90, λέει πρόεδρος, με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 με προφορική τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1. Υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έξι Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ. 7 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στη συνάδελφο κυρία Στρεβό, στους σκιώδες εισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε όλους. Νομίζω ότι πραγματικά με αυτές τις τροπολογίες βελτιώσατε πραγματικά το αρχικό μου κείμενο. Πρόκειται για μια έκθεση λοιπόν πραγματικά που αντικατοπτρίζει την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα στείλει με αυτήν την έκθεση ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ και εγώ πιστεύω ότι είναι ισχυρό μήνυμα αυτό που δίνουμε και για τις πολιτικές ε, της ε, νεολαίας. Ε, περιμένουμε και την έκθεση κομισιών αλλά και για τα θέματα εκπαίδευσης και τώρα περνάμε όπως είχαμε πει στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, Μόργανο και πάμε αμέσως ε, στις, ε, στην ψηφοφορία. Ελπίζω ότι έχετε όλοι το σχετικό δελτίο. Bene, cominciamo. Allora. Ξεκινούμε. Ένα, τροπολογία, ένα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 μάλλον 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 μίτσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 δεν ψηφίζουμε είναι γλωσσική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 δεν ψηφίζουμε για τον ίδιο λόγο. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψήφος 69 κατόπιν αιτήματος του Άλντε. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 χωριστή ψήφος ε, ζητούει το S&D πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές όχι ελέγχουμε. 78 ελέγχουμε. Oh. I close, sorry, I open the vote, I close the vote. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψήφο. 83. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89. Πάμε στην 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 92. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. 22 υπέρ, μία κατά, πέντε αποχές, συγχαρητήρια στον κύριο Μόργανο. Θέλετε να πείτε κάτι. Έχετε το λόγο. Ε, Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω θερμός ε, τους σκιώδεις ε, για την συνεργασία. Οι ευχαριστίες μου προφανώς και στην γραμματεία Κούλτ, στον κύριο Πόπα και όλους τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Είμαι πεπισμένος ότι η ομάδα της Επιτροπής μας βρίσκεται στην ενότητα των προθέσεών της πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλες ο πολιτικός αυτός στόχος επετεύχθη και αυτό διότι επεξεργαστήκαμε και τώρα διαβιβάζουμε στην Επιτροπή Τραν ένα μήνυμα σαφές και συνεπές με το οποίο υπογραμμίζουμε το ρόλο και τις δυνατότητες και τις προκλήσεις για να πάμε σε μια ε, πολιτική πολιτισμού βιώσιμη για τον, ε, τουριστικό, για τον πολιτιστικό τουρισμό το οποίο προσφέρει ένα μέσο για την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για τον τονισμό και την υπογράμμιση της ευρωπαϊκής ταυτότητας ε, που είναι πραγματική κοινωτήριος δύναμη συνολικά της οικονομικής μεγέθυνσης ε, των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ λέει η Πρόεδρος. Ήταν πράγματι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση αυτή. ήταν στην ουσία η πρώτη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου επί, του, επί θεμάτων τουρισμού και έχει εισαχθεί οριζόντια. Ευχαριστώ και εγώ τους ε, σκιώδεις και όλους που συνεργάστηκαν καθότι σε πέντε λεπτά θα καταφτάσουν οι εκπρόσωποι της Προεδρίας πραγματικά σας ζητώ το μεσημέρι ακριβώς να είμαστε εδώ για να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούν όλοι να είναι στην ώρα τους, ε, διότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είμαστε ακριβείς και να είμαστε στην ώρα μας. Θα πρέπει να διακόψουμε τώρα και να... Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε και να διακόψουμε Το διάλειμμα από ό,τι είχα καταλάβει ζητήθηκε για να μπορέσετε να συνεννοηθείτε και μεταξύ σας και ως σκιώδης και ως ε, εισηγητές. Το κάνατε ήδη δηλαδή μου λέτε. Γιατί η αναμονή είχε σχέση με αυτή τη δουλειά που έπρεπε να γίνει, τη συνεννόηση. Και εν πάση έχουμε ακόμα πέντε λεπτά. Chairman, η δυσκολία μου είναι ότι κάποιοι συνάδελφοι προσπάθησαν να είναι εδώ για να ψηφίσουν σε αυτή τη διάρκεια, σε αυτή την, το χρόνο που έχουμε αφιερώσει στην ψηφοφορία. Είναι εδώ δηλαδή για να συμμετάσχουν σε μία ψηφοφορία. Ήρθε κάποιος εδώ και είναι παρόν για να μπορέσει να ψηφίσει. Μπορούμε και τώρα να ξεκινήσουμε, αλλά πόσο, πόσο χρόνο έχουμε ακόμα μέχρι να έρθουν οι εκπρόσωποι. Σε δύο λεπτά θα έρθουν. Εντάξει, να ξεκινήσουμε άμα θέλετε. Συμφωνώ ότι υπάρχει εδώ μια σχετική σύγχυση. Είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε μια αναβολή της ψήφου, της ψηφοφορίας, για να μπορέσουν οι σκιώδεις, σε πάση περιπτώσει, να λάβουν γνώση και να συζητήσουν αυτά που σήμερα το βράδυ υπέβαλε η Επιτροπή. Τι να πω, μήπως πρέπει τώρα να γίνει η διαβούλευση, να βγουν έξω αυτοί που πρέπει να διαβουλευτούν εκτός της ε, αιθούσης, αλλά αυτό έχει νόημα από τη στιγμή που η Επιτροπή έχει υποβάλει κάποια πράγματα να τα λάβουμε υπόψη μας στην ψηφοφορία. Τι να σας πω, δεν θεωρείτε ότι πρέπει πρώτα να διαβουλευτούμε και μετά να ψηφίσουμε. Εν πάση περιπτώσει πριν έρθει η Προεδρία προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό πάντως να λάβουμε γνώση και να συζητήσουμε αυτά που υπέβαλε η Επιτροπή και να ψηφίσουμε στις 12. Μπορούν με αυτόν τον τρόπο οι σκιώδεις και οι συγγήτρια να συνεννοηθούν για το πώς θα ψηφίσουν. Ε, ναι, συμφωνώ διότι το αίτημα είχε νόημα πολιτικός. Δηλαδή ότι πρέπει να διαβλεφθούμε σχετικά με τις καινοτομίε τα νέα που προέκυψαν το βράδυ από τις περικοπές του Συμβουλίου κτλ. Αν είχαμε χρόνο πριν από την Προεδρία, αλλά δύο λεπτά δεν θα έφταναν, ήταν να σκεφτούμε από κοινού τι θα πούμε, δηλαδή να εξετάσουμε τα πιλωτικά κτλ. Και είχαμε συμφωνήσει ότι εφόσον είχαμε ανάγκη το χρόνο αυτό να ξεκινούσαμε τις 12 το μεσημέρι. Σδρογεύσκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, με τα χαράς να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τρία λεπτά θέλουμε μόνο. Έτσι ώστε... Διακόπτει ο πρόεδρος. Άρα λέει θα διακόψουμε όταν χρειάζεται για να επανέλθουμε τη ψηφοφορία. Κυρίε και κύριοι, αληθεύει ότι χθε το βράδυ περίπου στις 7 λάβαμε μία αξιολόγηση και δεν είχαμε πολύ χρόνο. Το προσωπικό μας έπρεπε να δουλεύει όλο το βράδυ και σήμερα το... θα έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε με μια μικρή αξιολόγηση. Έχει σημειωθεί μια πάρα πολύ μικρή βελτίωση και θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Έχουμε καταρχάς τα σημεία A, B, C και D. Εκεί θα λάβατε μια ιδέα με το, ε, για το τι έχει βελτιωθεί και τι όχι. σε περίπτωση που έχουμε A ή B, ε, προτείνω να ψηφίσουμε θετικά. Μετά, Υπάρχουν δύο περιπτώσεις για τις οποίες θα πρότεινα να μην ψηφίσουμε τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή Έκον και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προσπάθησα να καταρτήσω τον ακατάλογο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο προπολογισμό να μην χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία ήδη καλύπτονται από άλλους προπολογισμού, για παράδειγμα τον προπολογισμό υγείας ή οικονομικών. Μετά, προσπάθησα να δω τα ποσά που έχουν προταθεί στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε όταν ψηφίσει η Επιτροπή μας να εστιάσει καταρχάς την εκπαίδευση στον κινηματογράφο ε, υπάρχουν δύο προγράμματα σχετικά με τον υποτιτλισμό στην ε, τηλεόραση ή στον κινηματογράφο. Πιστεύω όμως πως είναι απόλυτα αναγκαίο να εστιάσουμε στα προγράμματα που καλύπτουν τη δημιουργικότητα, το Creative Europe και εάν δείτε κάποια αξιολόγηση στις συστάσεις, να σας υπενθυμίσω πως δεν υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις είναι προτάσεις που έχουν γίνει από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες κατόπιν εξέτασης των ποσών. Το σημαντικό είναι τα προγράμματα να συνεχίσουν, να μην διακοπούν για τον οποιονδήποτε λόγο. Υπήρξαν στο παρελθόν ορισμένες ε, περιπτώσεις με θετικές αξιολογήσεις και ορισμένες περιπτώσεις όπου προγράμματα διεκόπησαν. Το 2016 όμως πρέπει να φροντίσουμε να είναι καλύτερο από το 2015. Γι' αυτό πρέπει να αναφερθεί στην χρηματοδότηση. Σημαντικό είναι επίσης να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την σχέση ανάμεσα στις ε, πιστώσεις, πληρωμών και τις πιστώσεις αναλήψης υποχρεώσεων. Μετά, είναι ευκολότερο να εισαγάγουμε πιλωτικά προγράμματα με μικρότερο, χαμηλότερο προϋπολογισμό παρά πιλωτικά προγράμματα με μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Υπάρχουν κάποιες ε, συμβαστικές λύσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε αργότερα. Το σχέδιο, για το σχέδιο γνωμοδότησης της ε, Επιτροπής μας μπορούμε να έχουμε ένα ψήφισμα στο οποίο θα συμπεριληφθούν και κάποιες τροπολογίες της Επιτροπής ή κάποια σχόλια. Σίγουρα πρέπει να προστατεύσουμε την χρηματοδότηση για κάποια προγράμματα, για κάποιες ε, υποτροφίες, κάποιες επιχορηγήσεις ή προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ηθαγένεια και την ε, κατάρτιση. Όσον αφορά τροπολογίες για τον αθλητισμό πρέπει και αυτές να συμπεριληφθούν. Σας ευχαριστώ. Αν κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει εφόσον δεν έχουν καταφτάσει ακόμα οι πρόσωποι της Προεδρίας. Μόργανο. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα το πρωί έφτασε ένα αίτημα των Πρασίνων που έλεγε ας προσπαθήσουμε 5-10 λεπτά να συνεννοηθούμε εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σαν ομάδα να ψηφίσουμε αμέσως και δώσαμε και μία αξιολόγηση όταν το συναντηθήκαμε και το συζητήσαμε ότι συμφωνούμε να ψηφίσουμε εκείνα τα πιλωτικά με Α και Β και μετά επί τη βάση των πόρων θα κοιτούσαμε για κάποιες καινοτομίε που θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες. Μεταξύ των οποίων το, το προτινόμενο του συναδέλφου Διακόνου προκειμένου να δοθεί συνέχεια σε μια δουλειά που είχε ξεκινήσει και να μην διακοπεί. Τώρα εγώ ζητώ από τους συναδέλφους ε, των Πρασίνων ε, ποια είναι η πρόθεσή τους τελικά γιατί δεν ήταν κάτι για να αναβάλουμε αυτό που είχαν ζητήσει. Σε αυτή τη φάση λοιπόν τι λέτε να πάμε στην ψηφοφορία Μαραγκάλ. Πρόεδρε, έχοντας ακούσει τις εξηγήσει του συναδέλφου, νομίζω ότι μπορούμε να συμβήσουμε. Καταρχά την εντολή του εισηγητή, νομίζω, πρώτα, λέει η Πρόεδρος. Allora, prima di tutto noi voltiamo il mandato sul relatore per ripristinare... Πρώτα λοιπόν την ε, εντολή του συγγητή και μετά τις μεμονωμένες τροπολογίες επί του προϋπολογισμού. Διανάταση χειρός για την εντολή του εισηγητή για το γενικό προϋπολογισμό. Διανάταση χειρός υπέρ του να δοθεί εντολή. Μόνο για την εντολή λέω. Κατά. Αποχέ. Επομένω εγκρίνεται η εντολή προ τον εισηγητή. Για μένα καλύτερα να περιμένουμε την Προεδρία τώρα γιατί ξέρω εγώ. And then this. Allora, we try to vote and pray, uh, pray the presidency to, wait. If we are... Εντάξει, τότε θα κοιτάξουμε να ψηφίσουμε και θα ζητήσουμε από την Προεδρία να περιμένει. Γιατί φοβάμαι ότι μετά κάποιοι μπορεί να λείπουν και τα λοιπά. Τροπολογία ΚΑΛΤ 5801. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 02. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 03. Ε, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 04. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 05. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 07. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 06. Υπέρ. Όχι 04. 04. Μάλλον 4. Τώρα λέει η πρόεδρο. 08. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 09. <laughs> Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά απόχέ ελέγχουμε. Ε, close the Πέρασε. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε. Παρακαλώ. Για τη 15. Close the vote. Is... Απορρίπτεται απορρίπτεται. Υπέρ 16 ε, εγκρίνθηκε, 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 Uh, uh, close the vote. Rejected, sorry. 42 in favor. Το 42 τώρα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Το 42. Παρακαλώ. I close the vote. Πέρασε. Απορρίπτεται. Okay, this is this is done. Okay, this is the conclusion. Now we have not to to to go on. Okay, and so we are in time. The Λοιπόν, ωραία. Προλάβαμε. Η Προεδρία ήταν πολύ καλή μαζί μας. Τώρα θα υποδεχθούμε τους Υπουργούς. Καλωσορίζουμε την Προεδρία και σημαντικούς υπουργούς της κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, Κλοντ Μέντς, Υπουργός Παιδείας και Έρευνας, η κυρία Μάγκη Νάγκελ, Υπουργό Πολιτισμού. Θα συνεχίσω Ιταλικά. Θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα το πρωί, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε μαζί σας, γιατί φυσικά θέλουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να ενισχυθεί το πρόγραμμα για τον πολιτισμό και τους νέους Συνεχίζω λοιπόν στα Ιταλικά λέγοντας ότι θα κάνουμε ως εξή. Οι υπουργοί θα μιλήσουν διαδοχικά, πρώτα υπουργό Πολιτισμού και Τηλεοπτικών, Τηλεοπτικο-ακουστικών, μάλλον, και μετά θα έχουμε τον Υπουργό για θέματα παιδείας, μετά θα έχουμε παρεμβάσεις, απαντήσεις από τους ομιλητές, έχουμε περίπου μία ώρα και μισή. Και να πω τα εξή σύντομα μόνο ότι θεωρώ πως βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής σημαντικό για την Ευρώπη και λόγω της νέας ε, Προεδρίας Κομισιόν υπάρχει μια πιο πολιτική στρατηγική όθηση που εκτιμούμε αλλά βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε και μια ανησυχία που έχουμε ως Επιτροπή πολιτιστικών θεμάτων και εκπαιδευτικών και θεμάτων νεολαίας ότι στα 11 σημεία των πραγματικών προτεραιοτήτων δεν βλέπουμε τα θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Ως άξονες είτε νέας, νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου, κοινωνικού, και ξέρω ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου το έχει συμπεριλάβει αυτό ως άξονα, και δεν βλέπουμε επί των δύο αυτών θεματικών ε, κάποιους άξονες κινητικότητος ε, μεγέθυνσης οικονομικής και καλύτερης ε, απασχόλησης. Χωρίς διάσταση εκπαιδευτική και πολιτιστική η Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Το δείχνουν οι δυσκολίες τις οποίες διερχόμεθα και η χθεσινή πολύ δύσκολη ημέρα και το λέω και προς τους Έλληνες συναδέλφους όπου είχαμε μια σημαντική αποστολή στην Ελλάδα είχαμε προσπαθήσει να καταγράψουμε την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ακριβώς άξονα οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να επιταχύνει και να επανέλθει σε μια κατεύθυνση επενδύσεων επί των ανθρωπίνων πόρων, επί της κοινωνικής καινοτομίας και της πολιτιστικής καινοτομίας. Και ανησυχούμε διότι ακριβώς εχθές είχαμε την, ε, το νέο ότι το Συμβούλιο προέβλεψε κάποιες σημαντικές περικοπές του προϋπολογισμού. Εμείς μόλις ε, ψηφίσαμε τη γνωμοδέτηση του κυρίου Σντρογεύσκη, του εισηγητή μας, αλλά ακριβώς επί του θέματος της δημιουργικής πολιτικής και της ανακοίνωσης υπάρχουν στοιχεία λεπτομερείε που πάνε αντίθετα προς την στρατηγική μας αυτή προτεραιότητα. Εμείς λοιπόν ζητούμε από την Προεδρία να δεσμευθεί ε, για να αντισταθμίσει την κατάσταση αυτή. Και στο σχέδιο επενδύσεων Juncker είδαμε ότι αναφέρεται μεν η παιδεία, αλλά δεν είναι καθόλου σαφές με ποιο τρόπο προτείνονται χρηματοδοτήσεις. Και το Κοινοβούλιο ήταν που εισήγαγε τις ε, τον κλάδο της, ε, βιομηχανική, της ε, δημιουργικής με βιομηχανίας και της ε, εκπαίδευσης. Και θέλουμε να ακούσουμε τις προτεραιότητες του Λουξεμβούργου επί της πολυγλωσσίας, της πολιτικής για τους νέους και τα παιδιά και άλλων πολιτικών που θεωρούμε πολύ σημαντικές. Για τους νέους νομίζω ότι υπάρχει σημαντική δέσμευση της Βορειδίας. Εν πάση θεωρώ ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συνεργαστούμε καλά, αλλά σε αυτή τη σημαντική στιγμή σας ζητούμε να δώσετε ένα ισχυρό μήνυμα αλλαγής στην Ευρώπη, ώστε τα πολιτιστικά θέματα και εκπαιδευτικά να είναι πολύ περισσότερο εγγεγραμμένα στις προτεραιότητες και στην κατεύθυνση της πολιτικής. Θα δώσω τώρα μέσω το λόγο με μεγάλη χαρά στην ε, στον ε, Υπουργό Μάγκη Νάγκελ, στην Υπουργό Μάγκη Νάγκελ, συγγνώμη, για να μας παρουσιάσει ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε για την ε, υποδοχή σας και που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω πώς τους επόμενους έξι μήνες η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα βρεθεί στην υπηρεσία του πολιτισμού των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Δεν θα κάνω μία εισαγωγή όσον αφορά την αξία του πολιτισμού στην Ευρώπη, το ρόλο της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και το σεβασμό της πολυμορφίας στον τομέα του πολιτισμού. Πιστεύω ότι πρόκειται καθαρά για βασικές αξίες τις οποίες όλοι συμφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτή την αίθουσα. Και όλοι μοιραζόμαστε αυτή την πεποίθηση η οποία μας καθοδηγεί στην κοινή μας δράση προς όφελος του πολιτισμού και των ε, δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων. Δεν θέλω όμως να παραμείνω ασαφής και το άρθρο 167 της συνθήκης μας περιορίζει όσον αφορά αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε δυνατότητες, έχουμε περιθώρια λιγμών στους τομείς αυτούς και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για τον πολιτισμό. Τι θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, παρόλα αυτά που ακούγονται και παρόλη την κρίση, ο πολιτισμός παραμένει ουσιαστικός, γιατί ο πολιτισμός είναι καταρχήν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της συνύπαρξης, της συμβίωσης και ένα απόθεμα κοινών αξιών, κοινών σημείων αναφοράς, από τα οποία προκύπτουν συνειδήσεις, ε, κληρονομιές και φυσικά δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και πολλών άλλων. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να προσπαθούμε έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι το μέλλον της Ευρώπης περνάει σε μεγάλο βαθμό από τον πολιτισμό στους τρεις αυτούς τομείς που μόλις προανέφερα. Και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, γιατί είναι μεγάλη η συνεισφορά του πολιτισμού σε όλους τους τομείς για την ολοκλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην εθελοτυφλούμε. Σαν Υπουργοί Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουμε να επενδύουμε για να υπογραμμίσουμε τις θετικές επιπτώσεις αυτής της συνεισφοράς σε όλους τους δημιουργικούς τομείς του πολιτισμού συντονιζόμενοι με άλλους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής και προσπαθώντας να βρούμε συνοχή. Αυτό είναι μία πρόκληση και η Προεδρία του Λουξεμβούργου αποφάσισε να αναλάβει δράση ξεκινώντας από συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι θέλω να πω, θα μου πείτε, αφού σας ανακοίνωσα ότι δεν θέλω να είμαι αφηρημένη. Θα γίνω λοιπόν συγκεκριμένη. Σε σχέση με τους εταίρους μας, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στην κληρονομιά, στην οικονομική βιωσιμότητα και στην τεχνολογία και την καινοτομία, εμείς θέλουμε να βάλουμε το επίκεντρο της δράσης μας σε μια οριζόντια δράση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο τρίτος στόχος της ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την, τον πολιτισμό για την περίοδο 2015-2018. Επιθυμούμε λοιπόν να αναλάβουμε μια διαφορετική δράση. Σαν Λουξεμβούργοι είμαστε πιο ρεαλιστές και θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής. Στόχοι αναπτυξιακοί, λοιπόν, και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτον, πρόκειται για έναν τομέα όπου ο πολιτισμός έχει απτά αποτελέσματα και πολλά μπορούν να γίνουν στην πράξη με μία συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων, με καλύτερη διακυβέρνηση στον τομέα της μετανάστευσης της καλής ε, γειτονίας. Και βεβαίως το θέμα της ανάπτυξης, μία από τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή ε, Στρατηγική και η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Η ανάπτυξη όμως δεν μπορεί να είναι θέμα μίας ε, υπηρεσίας ή ενός τομέα. Τέταρτον, όσον αφορά τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η συζήτηση συνεχίζεται και βρισκόμαστε στην τελική φάση. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρούμε όμως ότι ο τομέας του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων αυτών. Τέλος, στόχοι και προγράμματα που έχουν προετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε σαν Συμβούλιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε για να το κάνουμε. Και πραγματικά τελευταίο σημείο, αλλά πολύ σημαντικό, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και τη δική σας εργασία, η έκθεση της κυρίας Ζάκα, αλλά και οι προτάσεις της Επιτροπής σας έχουν σαφώς θέσει πολύ σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, καθότι μπορεί η δική σας Επιτροπή να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ήπιας ε, δύναμης και από κοινού με τις προτάσεις της ε, Επιτροπής ε, Εξωτερικής Πολιτικής να παίξει το ρόλο της ενισχύοντας την πολιτιστική διπλωματία. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παίζει εδώ καθοριστικό ρόλο. Εχθές έγινε μια σημαντική ακρόαση εδώ στην Επιτροπή σας όσον αφορά την καταστροφή και την παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Γνωρίζουμε, το Συμβούλιο γνωρίζει τα προβλήματα αυτά και έγινε μια σημαντική συζήτηση τον προηγούμενο Μάιο. Υπογραμμίσατε τον επίγοντα κατά χαρακτήρα αυτής της καταστροφής. Αυτό το θέμα θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των σημείων που θέλουμε να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε. Θέλουμε λοιπόν εδώ πραγματικά να εκφράσουμε τη δέσμευσή μας και είμαστε πεπισμένοι ότι συνεργαζόμενοι μαζί σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με την Προεδρία μας θα μπορέσει να θέσει μια στεναρή βάση για να συνεχίσουμε την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και της πολιτιστικής διπλωματίας. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην συνάντηση που θα γίνει στο Λουξεμβούργο 3 και 4 Σεπτεμβρίου με θέμα πολιτισμός και ανάπτυξη για μια πιο στρατηγική προσέγγιση των πολιτικών στον τομέα του πολιτισμού και την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη Θέλουμε να δούμε πώς οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να ενισχυθούν από την πολιτική στο πολιτιστικό τομέα, ενισχύοντας τον ψηφιακό τομέα, τον πολιτιστικό τομέα και οι συζητήσεις αυτές θεωρούμε ότι σαφώς μπορεί να δημιουργήσουν μια νέα βάση για τη βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων και να δώσουν περισσότερη συνοχή και καλύτερη μεθοδολογία στη δράση μας. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπερασματικά θα πω ότι επικεντρωνόμενοι στον πολιτισμό θέλουμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη συνοχή στην πολιτική πολιτισμού, στην πολιτική ανάπτυξης και να υπογραμμίσουμε και την ανάγκη μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης του πολιτισμού και την ενσωμάτισή του στην εξωτερική δράση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα εργαλείο. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει και μπορεί να γίνει μέσω του πολιτισμού. Πρόκειται όμως πρώτα απ' όλα για μια αξία. Η πραγματική αξία του πολιτισμού ουσιαστικά βρίσκεται στις κοινωνίες που τους γέννησαν και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε όλοι μαζί στη συνειδητοποίηση ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μια θεμελιώδη αξία για το μέλλον και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για το πώς εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας σαν θα δώσω αμέσω το λόγο, κυρία Πρόεδρε, στο συνάδελφο και θέλω να πω και δύο λόγια ακόμα για τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά στον ψηφιακό τομέα. Αυτό βεβαίως δεν είναι δική μου αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια στρατηγική που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για το θέμα της ψηφιακής πολιτικής ένας τρόπος να διευκολύνουμε την οριζόντια ανάπτυξη. Ο ψηφιακός τομέας όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ξεχωριστός τομέας και οι θεσμοί στην Ευρώπη έχουν ε, ενισχύσει τις προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά στον ψηφιακό τομέα. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν εμπόδια για τις ε, υπηρεσίες που προσφέρονται online. Πρέπει να εξαφανιστούν αυτά τα εμπόδια για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να περάσουν τα σύνορα και να υπάρχει μια πραγματική πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα εθνικά ή άλλου είδους ε, προσκόμματα. Η πρώτη οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα ενισχύει τις ε, προσπάθειες της Επιτροπής να δημιουργηθεί στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων μία πραγματικά ελεύθερη κυκλοφορία. Η Προεδρία θα συνεχίσει να ενισχύει αυτή την προσπάθεια και βεβαίως περιμένουμε τα συμπεράσματα της Επιτροπής στο τέλος των διαβουλεύσεων για το θέμα της συζήτησης οδηγίας για τα οπτικά και τις υπηρεσίες στον τομέα αυτό. Η προσπάθεια λοιπόν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού τομέα στην Ευρώπη περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, εξυγχρονισμό των ε, κανόνων για τα πνευματικά δικαιώματα, για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου και βεβαίως περιμένουμε και νέες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της ε, Λουξεμβουριανής Προεδρίας. Θα προωθήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι η Επιτροπή για το 2016 θέλει να στηρίξει τις προσπάθειες για να δημιουργηθεί αυτός ο ενιαίος ψηφιακός κόσμος. Παρακολουθούμε με προσοχή αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα των online πλατφορμών, ιδιαίτερα για τον καθορισμό του περιεχομένου των οπτικοακουστικών μέσων με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής γι' αυτό και για τα άλλα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον τρόπο τον οποίο παρακολουθήσατε τις ε, εργασίες μας ως Επιτροπή έχουμε πολλές προτάσεις που μπορούμε να αξιολογήσουμε από κοινού, θεωρώ, ε, για στρατηγικές ε, επιλογές που πρέπει να γίνουν στο πεδίο αυτό. Ε, εκτιμώ και τη δέσμευσή σας σχετικά με την οδηγία και τις διαβουλεύσεις που τρέχουν. Θεωρώ ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε καλύτερη σαφήνεια συνολικά για τις προοπτικές που ανοίγονται για την συνολικά καλύτερη πρόσβαση αλλά και καλύτερο περιεχόμενο των πολιτιστικών ε, προγραμμάτων και πολιτικών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό Μένσου για τη δική του παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου για θέματα εκπαίδευσης νέων και μικρής ηλικίας. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τους ε, Ευρωπαίους ε, αυτή η δυνατότητα που μας δίνεται σήμερα να προωθήσουμε θέματα εκπαίδευση και καινοτομία. Όσον αφορά τι δικέ μα προτεραιότητε, η Προεδρία του Λουξεμβούργου είναι πεπισμένη ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε έμφαση σε μια ε, εκπαίδευση ποιοτική χωρίς αποκλεισμού για όλους τους νέους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε, να συμπληρώσουμε τις ε, εθνικές προσπάθειες με την ανταλογή βέλτιστων πρακτικών. Το 2009 τα κράτη-μέλη οφέτησαν το στρατηγικό πλαίσιο T 2020 με σκοπό να υπάρξει διάρθρωση της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού της εκπαίδευσης και το πλαίσιο αυτό αξιολογείται κάθε τρία χρόνια και παρουσιάζεται από κοινού με τις ε, πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτό βεβαίως ε, έγινε και με μια κοινή έκθεση Συμβουλίου και Επιτροπής και αυτό μέχρι το 2017. Το βασικό στοιχείο του προγράμματος της Προεδρίας θα παρουσιαστεί σε αυτά τα πλαίσια σαν μια κοινή έκθεση. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου βεβαίως θα κάνει έναν απολογισμό και θα καθορίσει τις προσπάθειες που πρέπει να συνεχιστούν από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου από τους νέους. Το θέμα αυτό των νέων που εγκαταλείπουν πολύ νωρί το σχολικό σύστημα είναι κάτι που βεβαίως γνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη και τα ποσοστά αυτών των νέων που πολύ νωρίς εγκαταλείπουν το χρονικό σύστημα είναι ανησυχητικά, ιδιαίτερα σε κάποιες κατηγορίες πολιτών όπως οι μετανάστες. Οργανώσαμε ένα συμπόσιο και φυσικά το Λουξεμβούργο θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια των συμπερασμάτων του συμποσίου αυτού για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Το θέμα επίσης της πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και της υποδοχής των μικρών παιδιών στο σχολικό σύστημα. Διαφορετικές πρακτικές θα πρέπει να ενσωματώσουν όλα τα παιδιά σε ένα πλαίσιο πολυμορφίας και πολυγνωσίας στο σχολικό σύστημα. Το Λουξεμβούργο οργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την εκπαίδευση μία ακρόαση με, θέα, με θέμα μία εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς, χωρίς αποκλεισμούς για τους νέους με σκοπό να δημιουργηθούν συμπεράσματα και προτάσεις για μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς περιορισμούς και να προετοιμάσει μία ευρωπαϊκή ατζέντα μέσω της οποίας όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι νέοι θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι ώστε να δούμε και το θέμα της απασχολησμότητας των νέων, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, κάτι που θα πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας και να συμπεριλάβει νέους κάθε κοινωνικής κατηγορίας με σκοπό να προωθήσουμε την πολυμορφία και την πολυγνωσία των νέων πολιτών της Ευρώπης, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα κυρίως από τότε που 28 υπουργοί το Μάρτιο του 2015 το υπογράμμισαν στη δήλωση του Παρισιού. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η στιγμή που αναλαμβάνουμε την Προεδρία μας, καθότι ξεκινάμε το δεύτερο κύκλο του προγράμματος 2010-2018, οργανώνοντας περαιτέρω τον διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των νέων της Ευρώπης και ολοκληρώνουμε την δεύτερη φάση των εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους νέους. Αυτό θα αποτελέσει βεβαίως βάση για περαιτέρω συζήτηση και σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης. Θα προτείνουμε λοιπόν στο Συμβούλιο ένα ψήφισμα, μια έκθεση για το θέμα αυτό που θα βασίζεται στο διαρθρωμένο διάλογο για θέματα νέων. Στο Συμβούλιο του 2015 οι Υπουργοί πολιτισμού και νεότητας στη Ρήγα το Μάρτιο του 2015 έβαλαν ειδική προτεραιότητα στο θέμα της συμμετοχής των νέων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και από τις 21-24 Σεπτεμβρίου στην συνδιάσκεψη που οργανώνουμε στο Λουξεμβούργο και με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε προσκεκλημένους και συμμετέχοντες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ολοκληρωθεί ο τελευταίος διάλογος αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου με σκοπό να φτάσουμε σε τελικά συμπεράσματα τα οποία τελικά θα υποβληθούν στους υπουργού Νεότητας το Νοέμβριο του 2015 στο Συμβούλιο Υπουργών. Η Προεδρία θέλει επίσης να εξετήσει για το 2015 μια κοινή έκθεση για θέματα νέων, μια μεσοπρόθεσμη έκθεση, έναν απολογισμό για τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα νέων. Τέλος, θα προτείνουμε να υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα για δράση προς όφελος των νέων, προτείνοντας τις μεγάλες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2016-2018. Από τη μία θα πρόκειται για δράσεις, για περισσότερα προγράμματα σε επίπεδο εκπαιδευτικό και κοινωνικό και την στήριξη νέων όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης. Επίσης, σημαντική θέση κατέχει η προσπάθεια εξάλληψης του αποκλεισμού, της αποδέσμευσης και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων να βοηθήσουμε το πέρασμα των νέων στην ε, ενήλικη ζωή και στην εξέβρεση θέσης απασχόλησης. Επίσης, θέματα που άπτονται της υγείας και της ευημερία των νέων, οι νέες αυτές πολιτικές προσφέρονται στους νέους και στον ψηφιακό κόσμο στον οποίο κινούνται σήμερα. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη μας και το σχέδιο Juncker και όλες τις δυνατότητες να ενσωματώσουμε στοιχεία στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων, σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει βεβαίως να καθοριστεί ο τύπος των προγραμμάτων που θα στηριχτεί μέσω αυτών των κονδυλίων, πέραν δηλαδή του σχεδίου Juncker για τους νέους και την παιδεία. Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε προτάσεις για την ανάπτυξη των πολιτών, κυρίως όμως για την κατάρτιση των νέων, για να τους δώσουμε νέες προοπτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για την πρόσκλησή σας, για την προσοχή σας και για το ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πρόγραμμα εργασιών και τις πρωτοβουλίες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Με χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας και θα δεχτώ τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Τον ευχαριστούμε θερμός. Έχουμε πολύ καλές βάσεις για την κοινή μας δουλειά. Μας ενδιαφέρει η έκθεση για τους νέους στην οποία αναφερθήκατε και το γεγονό ότι θέλετε να δώσετε μια προσοχή πιο ενδελεχή, πιο λεπτομερή στο σχέδιο Juncker σε ό,τι αφορά τις θεματικές αυτές και εμείς ε, μόλις ε, εγκρίναμε μια γνωμοδότηση για την εκπαίδευση και την ε, επιχειρηματικότητα των νέων ακριβώς σήμερα και είχαμε και μια σημαντική γνωμοδότηση της συναδέλφου Ριμπάτσκα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπρόνια όπου είχαμε και το συνέδριο το διετές ε, φέτος <clears throat> για να καταλάβουμε τις προοπτικές ε, των πολιτικών εκπαίδευσης ή στην Ευρώπη. Τώρα, έχω εγγράψει κάποιους... Ε, Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε κυρίες Υπουργοί, για την παρουσίαση των κύριων σημείων της, του προγράμματος της δικής σας Προεδρίας. Ένα ερώτημα μου δημιουργείται αυτή εξ αρχής. Έχουμε συζητήσει για τον προπολογισμό εδώ στην Επιτροπή και διαπιστώνω ότι ακριβώς στα, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες έχει γίνει πρόταση από την ε, Επιτροπή να περικοπεί ο προπολογισμό τα επόμενα χρόνια και αυτό μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση διότι από τη μία θέλουμε να προωθήσουμε τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και πρέπει να αποφύγουμε να βγάζουμε τα κονδύλια από κάπου και να τα ε, δίνουμε κάπου αλλού. Πιστεύω πως ε, δεν θα προχωρήσουμε ε, και δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας να προωθήσουμε την κατάρτιση, να αυξηθεί η κατάρτιση και απασχοληθμοσιμότητα στους νέους αν γίνονται περικοπές. Γι' αυτό λοιπόν θα Ήθελα να σας τονίσω πως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν περικοπές στον τομέα της ε, εκπαίδευσης της, ε, των νέων. Χρειάζονται κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να προέλθουν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ε, και χρειάζεται ενίσχυση ίσως από εκεί. Διαφορετικά δεν μπορώ να πω ότι προβλέπω να έχουμε πρόοδο σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται προσοχή και από τη δική σας Προεδρία και από τις επόμενες. Τώρα, σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά. Πιστεύω πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα από την ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει και προηγουμένως στην συζήτηση για το πακέτο των ε, τηλεπικοινωνιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί και ο τομέας του πολιτισμού, να υπάρχουν πολλές δυνατότητες στην ψηφιοποίηση η ψηφιοποίηση μάλλον πρέπει να συμπεριληφθεί η πολιτισμική πολυμορφία, η ελευθερία Απόψη η ουδετερότητα του διαδικτύου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια της ψηφιακή ενία αγορά. και αυτά τα θέματα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τον πολιτισμό. Θα ήθελα ε, λοιπόν να δω κάποια μεγαλύτερη πρόθεση ενασχόληση από την Προεδρία σας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κάμερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε, κυρία Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ απόλυτα με την προλελή σας, την Σαμπίνα Φερχάιεν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαμε πολλές έντονες συζητήσεις, πολεμήσαμε για να κρατήσουμε το πρόγραμμα Erasmus+. Όμως, από όλες τις εθνικές αρχές και υπηρεσίες μαθαίνουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή. Ιδιαίτερα στην εφαρμογή του προγράμματος για τους νέους, οι οποίοι μας απασχολούν ιδιαίτερα ως Επιτροπή Πολιτισμού. Θέλουμε να στηρίξουμε το κοινωνικό κεφάλαιο, τους ε, νέους, και από ό,τι μαθαίνουμε ο τομέας της άτυπης ε, κυρίως κατάρτισης των μικρών προγραμμάτων πάσχει. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή, σοβαρές δυσκολίες και μάλιστα το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από το επιθυμητό. Τα μικρά, μικρής έκτασης προγράμματα δεν στηρίζονται. Αυτό το βλέπουμε και στο πρόγραμμα Λεωνάρτο Νταβίντσι, όπου έχει παρατηρηθεί πως λείπουν οι θεσμικές δομές έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ε, νέους αποφύτους να κάνουν πρακτική σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Όλες αυτές λοιπόν οι δυσκολίες και τα προβλήματα στην εφαρμογή απειλούν την επιτυχία του προγράμματος και πάντα λέγαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή η οποία αυτή τη στιγμή είναι κάθε άλλο παρά καλή. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να δώσετε λίγη περισσότερη βάση στον ε, τομέα αυτό. Μάλιστα εν ώψη και της ενδιάμεσης αναθεώρησης που θα γίνει σε λίγο καιρό. Χρειάζεται μαζί Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα αυτό και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Ε, τώρα, Όσον αφορά την πολυγλωσία, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίασή σας. Έχουμε παρατηρήσει ότι έχει ανοίξει μια νέα συζήτηση σε πολλά κράτη-μέλη σχετικά με την ενίσχυση της πολυγλωσσίας, ιδιαίτερα ε, σχετικά με τις αποφάσεις κάποιων κρατών να περιορίσουν τα γλωσσικά μαθήματα της Γαλλίας, για παράδειγμα, που περιόρισε τη διδασκαλία των γερμανικών στα γαλλικά σχολεία. δίδεται περισσότερη βάση στα αγγλικά. Χρειάζεται όμως να προωθηθούν και άλλες γλώσσες. Πιστεύω πως είναι κάτι αρκετά σημαντικό, το οποίο έχετε παρουσιάσει ως προτεραιότητα και στα πλαίσια της, ε, του ψηφιακού θεματολογίου θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με την ΕΣΑ Φερχάιεν και να την στηρίξω. Να προσθέσω επίσης το θέμα του, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιμένω να ακούσω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτό. Θεωρώ όμως πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να βρεθεί η σωστή ε, ισορροπία στην πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά. Ακούμε πολύ συχνά ότι πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να αμείβονται επαρκώς για το έργο τους, όμως από την άλλη πρέπει να προσέξουμε επίσης και η πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά να είναι εύκολη. Χρειάζονται κανόνες και κανόνες για εξαιρέσεις ε, ορισμένων πολιτισμικών αγαθών. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός δεν δημιουργείται μόνο, αλλά υπάρχει και ε, διαθέσιμος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε όχι μόνο για την δημιουργία πολιτισμικών αγαθών, αλλά και για την πρόσβαση στα ήδη φυστάμενα πολιτισμικά αγαθά. Χρειάζεται, όπως είπα, ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργία και στην διατήρηση και στην πρόσβαση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως Προεδρία του Συμβουλίου έχετε κάποια ε, συγκεκριμένη πρόταση, δίδετε κάποια έμφαση και επίσης σας μην ξεχνάμε και τον γεωγραφικό περιορισμό, το geo-blocking, το οποίο ε, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Εσείς ως Προεδρία πόσο σκοπεύετε να δράσετε. γιατί αυτό πρέπει να συζητηθεί και σε συνδυασμό με την ε, προσβασιμότητα και με την φορητότητα. Και περιπλέκεται επίσης το θέμα, διότι τα πνευματικά ε, δικαιώματα δεν αφορούν μόνο το διαδίκτυο, αλλά και την ραδιοτηλεόραση Έχω για παράδειγμα κατά νου διεθνείς άδειες, πανευρωπαϊκές άδειες για συγκεκριμένα οπτικοακουστικά μέσα. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί, διότι θα ωφελήσει μόνο τις, ε, τους πολυεθνικούς ομίλους, ιδιαίτερα ε, εκείνους που εδράζουν στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα λειτουργήσει αρνητικά για τους ε, μικρότερους παρόχους των ευρωπαϊκών κρατών. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι γίνεται σχετικά με την κατάργηση των ε, γεωγραφικών περιορισμών. Εκεί φαντάζομαι πως θα συναντήσετε περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή παρά στο ζήτημα της εφορητότητας. Η κυρία Τρουπελ. σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω τα όσα είπαν οι προλελήσεις σας, η κυρία Φερχάριν και η κυρία Κάμερεβερτ. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον ε, γεωγραφικό ε, αποκλεισμό. Διότι διακυβεύεται και η πολιτισμική πολυμορφία. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία. Ε, τώρα, όσον αφορά τις ε, πολιτισμικές εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, είναι απόλυτα αναγκαίο, όπως έχουμε ήδη ε, συζητήσει, να μην κοιτάζουμε από πάνω προς τα κάτω, αλλά να δραστηριοποιηθούμε από τη βάση με διάφορες πολιτισμικές ε, παρεμβάσεις όταν αυξάνονται οι εντάσεις ε, ορισμένα μέλη. Θα ήταν ίσως καλό να έχουμε κάποια κονδύλια έτσι ώστε να, σε τέτοιες περιπτώσεις να διευκολύνεται ο διάλογος για την εξομάλυνση των ε, εντάσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν έχετε πρόθεση να εφαρμόσετε κάτι τέτοιο και επίσης να σας ρωτήσω για το τι γίνεται με το Erasmus Plus. Τώρα, συζητήθηκε επίσης ότι στο πρόγραμμα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση παρατηρήθηκε μία τάση να προτιμώνται τα μεγαλύτερα προγράμματα. Μας υποσχέθηκαν πως θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος, ιδιαίτερα στα σχολεία πώς θα δίδεται βάση στα μικρότερα προγράμματα που θα στηρίζουν τον πολιτισμό. Ε, είστε λοιπόν έτοιμοι να ακολουθήσετε αυτήν την γραμμή, να δημιουργηθεί κάποια εκτελεστική αρχή που θα επιβλέπει έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εφαρμογή μικρών πολιτισμικών προγραμμάτων. Ο έχει το λόγο. Ο ε, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, ε, αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ε, και είναι χαρακτηριστικό ότι πέραν από τα μεγάλα λόγια για τον πολιτισμό που ακούμε συνέχεια, ή θα έλεγα οι δαπάνες συνεχώς μειώνται και τα προβλήματα στον πολιτισμό αλλά και στην παιδεία πολλαπλασιάζονται. Σας εύχομαι λοιπόν πρώτα απ' όλα καλό κουράγιο και με ικανοποίησε ότι έχετε μια πιο συγκεκριμένη, θα έλεγα, αντίληψη των πραγμάτων. Θέλετε να αφήσετε συγκεκριμένα ίχνη κατά την παρουσία σας ε, το σημαντικό αυτό εξάμεινο από όπου όπως ξέρετε ακόμα και η ιδέα της Ευρώπης που συνένωσε πολλούς λαούς αφισβητείται από πολλές πλευρές. Έτσι το έργο σας στον πολιτισμό και στην παιδεία γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Για μας τους Έλληνες ήταν μια πικρή εμπειρία ότι δοκιμάστηκε ακόμα και η, θα έλεγα η έξοδος της Ελλάδα από την Ευρώπη δοκιμάστηκε, ευτυχώς για την ώρα τα πράγματα ηρέμησαν το ότι μόνο τέτοιες σκέψεις υπάρχουν από πολλές πλευρές νομίζω ότι δείχνει ότι ο πολιτισμός είναι και αυτό σε κρίση γιατί αν μη τι άλλο η Ελλάδα όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα μακρόχρονο και πολύ σημαντικό πολιτισμό και ιδεώδη δημοκρατικά. Δεν θέλω λοιπόν να σας κάνω πολλές ερωτήσεις. Να επαναλάβω μόνο και εκεί θα ήθελα και εγώ μια περισσότερο συγκεκριμένη απάντηση ότι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί αναζητείται μια ισορροπία δύσκολη, πολλές φορές επικίνδυνη και ακόμα και αυτή η Επιτροπή εδώ του πολιτισμού παρά τις καλές της προθέσεις ε, απέτυχε να εκφράσει μια ολοκληρωμένη πρόταση γύρω από τα δικαιώματα των πολιτεχνών γύρω από τα φοβερά προβλήματα που παρουσιάζονται, πράγμα που ήταν μια μεγάλη απογοήτευση για μένα. Ελπίζω λοιπόν ότι εσείς θα προχωρήσετε τουλάχιστον 3, 5, 6 μικρά βήματα. Ας μην μείνουμε όμως στη στασιμότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έδινα τώρα το λόγο για τις απαντήσεις σας. Δεν βλέπω άλλους συναδέλφους να ζητούν το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ την Υπουργό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επανέλθω στην τοποθέτηση της κυρίας δερούβεν ε, για την ε, κοινή αγορά, την ψηφιακή ε, και έχετε απόλυτο δίκαιο. Είναι δυστυχές ότι είχαμε περικοπές ιδιαίτερα τα διατομεακά και τα πολιτιστικά του προϋπολογισμού και πολύ συχνά βλέπουμε δυστυχώς ότι τα πολιτιστικά είναι αυτά που θυσιάζονται πρώτα. Αυτό συνδέεται με αυτά που σας έλεγα νωρίτερα για την φήμη συνολικά που θα μπορούσαμε να έχουμε στον τομέα του πολιτισμού. Ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ε, για τη διατομεαγότητα και τον οριζόντιο χαρακτήρα των πολιτικών πολιτισμού. Και δεν έχουμε επιλογή. Και πρέπει να ε, λαμβάνουμε υπόψη μας και δύο ακόμα στοιχεία σχετικά με την τοποθέτηση του Συμβουλίου. Γνωρίζουμε ότι τα δημοσιονομικά στην Ευρώπη είναι ακόμα υπό τη σκιά της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσεως και της επίπτωσης που αυτή η τελευταία είχε πάνω στον προπολογισμό. Ε, κατανοούμε το ρεαλισμό που πρέπει να έχει το Συμβούλιο για τα δημόσια οικονομικά, αλλά έχουμε ακόμα μεγαλύτερες περικοπές. Ε, έχουμε μάλλον λίγο μεγαλύτερο προϋπολογισμό από εκείνον του 2015 για το αντίστοιχο πρόγραμμα των δημιουργικών πολιτικών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά το υλικό αυτό κατά τη διάρκεια και θα το κάνουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας μας. Εμείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην, στο πρόγραμμα Creative Europe και ως προς την πρόθεση των ε, ταμείων των μέσων χρηματοδότησης αυτών των πολιτικών ε, ελπίζω να έχουμε ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο ε, για την ψηφιοποίηση αυτό είναι κάτι συνεχές στο θεματολόγιο του Συμβουλίου που εδώ και πολλά χρόνια έχει σχηματίσει ένα, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών η οποία θα δημοσιεύσει την επόμενη έκθεσή της στο φθινόπωρο. Εμείς ε, θα τη χρησιμοποιήσουμε, έχουμε κάθε πρόθεση να το κάνουμε, ε, μένει στο κέντρο των ανησυχιών μας ε, και ως προς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά και ως προς τα βιωσιμότητα. Για την κυρία Καμρέβετς αυτά που είπατε δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συμπεριλάβουμε την, το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού, να αναδείξουμε τη σημασία του και να βρούμε μία φωνή και μία κατεύθυνση θα έλεγα σαφή και συνεπή μαζί με τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Γραμματικάκη να πω ότι βεβαίως και γνωρίζουμε, αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πλήρως. Έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε έτσι όπως είπατε με μικρά βήματα προς τα εμπρός, αλλά είμαστε απόλυτος πεπισμένοι ε, για την κατεύθυνση που, θα, που θέλουμε να ακολουθήσουμε σε αυτά τα μικρά βήματα και για τα θέματα πολιτισμού και για τα θέματα βεβαίως παιδείας. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μένς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα γερμανικά για τις ε, ε κυρίες ε, που με ρώτησαν στα γερμανικά. Κύριε Φερχάιεν, έχετε εκφράσει κάποιους φόβους σχετικά με το ότι υπάρχει ο κίνδυνος να παίρνουμε κονδύλια από ένα ταμείο, να τα πηγαίνουμε στο άλλο και να το πουλάμε αυτό ως ε, επιτυχία. Πιστεύω πως η Προεδρία μας θα είναι, σε, θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική και θα είναι πάντα επάγνυπνη χρειάζεται προσοχή στις επενδύσεις. Πρέπει να γίνονται σωστές επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού. Και δεν ε, αρκεί μόνο να επενδύονται κονδύλια, χρειάζεται και η σωστή πολιτική και τα σωστά κίνητρα για να πραγματοποιηθεί αυτή η πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή, σωστές επενδύσεις, σωστά κίνητρα έτσι ώστε το σχέδιο Juncker να ωφελήσει τους νέους, να ωφελήσει τον πολιτισμό. Το δικό μας πρόγραμμα είναι λίγο πολύ εναρμονισμένο με το πρόγραμμα Juncker. Χρειάζεται η δημιουργία μόχλευσης και αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο με, την, ε, με τις επενδύσεις στις, στις νέες τεχνολογίες, στους νέους. Και πρέπει αυτή, αυτός ο διάλογος να λάβει χώρα όχι μόνο μεταξύ ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, αλλά και να συμπεριληφθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται συνεργασία λοιπόν όλων των ε, θεσμικών οργάνων και των ε, κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους ε, στόχους της Προεδρίας μας και τους στόχους του σχεδίου Juncker. Κυρία Καμερέβερτ, αναφερθήκατε επίσης σε ένα πρόβλημα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+. και αναφερθήκατε στην ευθύνη τόσο της πολιτικής όσο και του ε, διοικητικού τομέα. Αναφερθήκατε στην έλλειψη θέλησης εφαρμογής της θεωρίας. Να σας πω ότι καμιά φορά είναι προς όφελός μας ε, το ότι είμαστε πολιτικοί σε μια μικρή χώρα και μπορούμε να επιβλέπουμε καλύτερα το τι γίνεται σχετικά με την εφαρμογή εκεί. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αμέσως εάν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην εφαρμογή του Erasmus Plus και να αντιδράσουμε άμεσα λοιπόν. Μας είπατε επίσης πως ε, είναι γεγονός ότι τα μικρά προγράμματα δεν προωθούνται και δεν στηρίζονται. Προγράμματα που στηρίζουν όχι μόνο την τυπική εκπαίδευση αλλά και την άτυπη, άτυπη κατάρτιση. Χρειάζεται να κάνουμε μία ανάλυση, είναι η απάντησή μου, για να εντοπίσουμε ποιοι τομείς ε, να εντοπίσουμε τους τομείς οι οποίοι χρειάζονται απλούστευση και εκείνους που χρειάζονται βελτίωση και να κάνουμε τις προτάσεις μας. Αναφερθήκατε επίσης στην γερμανική ε, γλώσσα και την προώθηση της. Πιστεύω πως ε, δεν είναι μια αρμοδιότητα της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε στο γενικότερο πλαίσιο της επικουρικότητας και της εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει φυσικά τις δικές της προτεραιότητες και, θα, και καλώς τις έχει, τη δική της ταυτότητα, τον δικών της ε, πολιτισμό και αυτό αφορά και την γλωσσική πολυμορφία μιας χώρας. Φυσικά βέβαια η Προεδρία μας θα προσπαθήσει να τονίσει την σημασία της πολυγλωσσίας. Της πολυγλωσσίας σε μια μεγάλη Ευρώπη η οποία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τις εθνικές ταυτότητες αλλά και από την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Την ευρωπαϊκή ταυτότητα σε αντιπαράθεση με την ε, παγκόσμια. Σίγουρα η γνώση περισσότερων γλωσσών είναι προς ωφελός μας όταν μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερους πολίτες στη δική τους γλώσσα, να συνεννοηθούμε με περισσότερους πολίτες στη δική τους γλώσσα. Σίγουρα η γνώση περισσότερων γλωσσών μας δίνει και καλύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό μιας ε, χώρας και σε καλύτερο διάλογο. Είμαι σίγουρος πως η πολυγλωσσία θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν διαβάζει κανείς τις επιστημονικές και στατιστικές μελέτες που δείχνουν ότι η εκμάθηση γλωσσών αυξάνει την ε, ευφυΐα, μειώνει το ενδεχόμενο εμφάνισης ε, μορφών άνοιας αργότερα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προωθείται η πολυγλωσία από μικρή ηλικία, από παιδική ηλικία. Η δική μας εμπειρία είναι χαρακτηριστική. Είμαστε μια χώρα με πάρα πολύ λίγους κατοίκους. Η μισή από αυτούς μιλούν Λουξεμβουργιανά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες έτσι να, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους γειτονές μας. τον κύριο Γραμματικά θέλω να ο οποίος επέμεινε πολύ στην σημασία των επενδύσεων στο πεδίο της παιδείας, της εκπαίδευσης και είχε, αν θα μπορούσα να πω, μια πισιοδοξία στην τοποθέτησή του. Προφανώς ε, ο καθένας βιώνει την πραγματικότητα στο πλαίσιο της χώρας του, αλλά έχουμε και μια συνολική ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Εγώ δεν δεν θα ήθελα να είμαι τόσο απεσιόδοξο. Γιατί νομίζω ότι έχουμε καταλάβει στην Ευρώπη ότι ε, αν θέλουμε να αναπτύξουμε την Ήπειρο αυτή, να προετοιμάσουμε το μέλλον μας, αν, έχουμε, αν θέλουμε να έχουμε και ακόμα και οικονομική επιτυχία, πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους, πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία, στην κατάρτιση των νέων, για να τους δώσουμε τα εργαλεία, τα μέσα που θα χρειάζονται σε 20-30 χρόνια ώστε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Χρειάζονται λοιπόν ε, χρειάζεται η ανάπτυξη των προσωπικών εκείνων δεξιοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας, το αυτό είναι προφανές, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων ε, της ε, οικονομικής ζωής, αλλά και στην ιδιωτική της ζωή, αλλά πρέπει να τους προετοιμάσουμε και ως υπεύθυνου πολίτες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν σε ένα δημοκρατικό διάλογο, να δεσμεύονται, να υποστηρίζουν ε, τις αξίες της δημοκρατίας. Και μέσω της επαφή που έχω καθημερινά με γονείς, με μαθητές ε, σχολικών ιδρυμάτων, ε, νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι απολύτως κατανοητό. Στη χώρα μου τουλάχιστον, αλλά είμαι βέβαιος και σε όλες τις άλλες χώρες. Βεβαίως και διερχόμεθα μιας φάσης εξαιρετικά σοβαρής, κρίσιμης για τα θέματα προϋπολογισμού, για πολλά δημοσιονομικά θέματα πολλών κρατών μελών και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, να δίνουμε την κατάλληλη εκπαίδευση στους ε, μελλοντικού μας πολίτες και να μην έχουμε υπερβολικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των πολιτικών παιδείας. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος για την παρέμβασή σας αυτή. Βλέπω την κυρία Τρούπολ, δεν ξέρω αν και άλλοι συνάδελφοι θέλουν και πάλι το λόγο. Ε, παρακαλώ. Και ο κύριος Δρογεύσκη. Έπρεπε να βγω για δύο λεπτά και δεν μπορούσα να ακούσω την αρχή της τοποθέτησής σας. Αλλά ήθελα να πω σχετικά με αυτό το πιθανό, το δυνητικό ε, ταμείο παρέμβασης για τα θέματα πολιτισμού, όπως και για το μικρότερο πρόγραμμα. Ήθελα να καταλάβω αν το παρακολουθείτε αυτό και αν θα κάνετε κάποια, και κάποιο follow-up, κάποια δράση μετά από... Μάλλον για να παρακολουθήσετε καλύτερα την εξέλιξη αυτή. Ο κύριος Σεσδρουγεύσκη. Ε, πρόεδρε, θα αναφερθώ σε κάτι που έχει αποσχολήσει όλες τις προηγούμενες προεδρίες που έχουμε βιώσει, τα στατιστικά στοιχεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση και γνώση για τα θέματα προϋπολογισμού, για τις δαπάνες δηλαδή των κρατών μελών, για θέματα πολιτισμού και παιδείας. Για παράδειγμα, για τη χρηματοδότηση ε, μεμονωμένων προσπαθειών ε, κινηματογράφου για παράδειγμα, παραγωγών κινηματογραφικών. Αν δούμε τις ε, πολιτιστικές ε, δαπάνες για παράδειγμα στη Γερμανία και στη Γαλλία, τότε η κατηγοριοποίηση των δαπανών στον προϋπολογισμό είναι τελείως διαφορετική μεταξύ τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθορίσει κανείς πόσο σημαντικά είναι τα θέματα πολιτισμού για την κάθε χώρα επί τη βάση του προϋπολογισμού και των κονδυλίων έτσι όπως καταχωρίζονται στον ε, προπολογισμό. Δεν ξέρω αν η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα κάνει μια προσπάθεια εναρμόνισης αυτών των ε, μέτρων ώστε να κατανοούμε καλύτερα τι δαπανούμε τελικά για τα θέματα πολιτισμού. Παρακαλώ την κυρία Evans. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά άκουσα την έμφαση που δίνεται στην πολυγλωσία. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία που είναι δίγλωση χώρα και δίδουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη χρησιμοποίηση των Ουαλικών μαζί με τα Αγγλικά που τα ομιλεί η πλειοψηφία. Αλλά τα περισσότερα θέματα πολιτισμού είναι στην αρμοδιότητα της ουαλικής κυβέρνησης. Και ήθελα να καταλάβω κατά πόσον θα υπάρχει ενεργός ε, συνεργασία όχι μόνο με τις κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και με τις περιφερειακές ημιαυτόνομες κυβερνήσεις για την υλοποίηση θεμάτων πολιτισμού και εκπαιδευτικών θεμάτων. Έχουμε άλλους, ε, άλλες ερωτήσεις? Όχι. Από βλέπω, όχι. Θα προσθέσω και εγώ δύο ερωτήματα Καταρχάς να σας πω ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος ε, και η πρόκληση συνολικά στο εκπαιδευτικό για τα θέματα ακριβώς ε, διαπολιτισμικότητας ε, θα έχουμε και μια ακρόαση το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή μας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της UNESCO διότι θα έχουμε και την, τα 10 έτη από τη σύμβαση του UNESCO για την παγκοσμιότητα την πολιτιστική. Επομένως θα ήθελα να τονίσω να υπογραμμίσω και αυτή τη διάσταση για τα θέματα τα εκπαιδευτικά και τα πολιτισμικά και νομίζω και εδώ θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας και για την ε, πολυγλωσία. Είναι αλήθεια ότι αυτό από τα κράτη-μέλη. Αλλά όπως έλεγε και η κυρία Κάμερεβερ, οι πρόσφατες ε, τροποποιήσεις που έχουν γίνει εθνικά δεν πηγαίνουν προς την ε, κατεύθυνση των συστάσεων των ευρωπαϊκών που συνιστούν μία μητρική και δύο ξένες γλώσσες στους κύκλους σπουδών. Κινδυνεύουμε, λέει ο να πάμε σε μία μόνο ξένη γλώσσα στους κύκλους σπουδών. Μόνο μία. Και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ενισχύσουμε, μάλλον να αντισταθμίσουμε το γεγονός αυτό, θυμίζοντας το πλαίσιο των ε, συστάσεων που είχαν δοθεί για τη συνεργασία στο πεδίο αυτό. Το άλλο <clears throat> που ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είμαι βέβαιο ότι τελικά θα έχει έτσι, για το συνέδριο επί της έκθεσης ε, ε, για τους νέους και για τα πρόγραμμα Erasmus Plus που είχαμε μια πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν και μετά ευτυχώς το Συμβούλιο δεν περιέκοψε και πάρα πολύ διατηρήθηκε ένα κάποιο επίπεδο χρηματοδότησης, όπως και η συνέπεια επί των προγραμμάτων για τους νέους κυρίως. Ήθελα λοιπόν απλώς να, επαληθευ... να επιβεβαιώσετε αυτά αν μπορείτε. Εμείς επίσης να σας πω μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η, η πολιτιστική διπλωματία αν θέλετε δηλαδή η εξωτερική πτυχή για να το πω έτσι της πολιτιστικής ε, ε, πολιτικής ε, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που έχουμε και σε θέματα γειτονίας επομένως είτε η Creative Europe είτε οι πολιτικές για τους νέους θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι συμπεριλαμβάνουν ένα, μία πτυχή εξωτερικής διαστάσεως και διαστάσεως γειτονίας γιατί νομίζω ότι είναι όλο και πιο απαιτούμενο και φαντάζομαι και ελπίζω ότι στις διμερείς επαφές που θα, στις οποίες θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλαμβάνεται αυτή η πτυχή που περιλαμβάνεται στο Erasmus μόντους. Ε, παρακαλώ τώρα για την ε, τελευταία σας ε, παρέμβαση ε, πρώτα τον Υπουργό Μέλσο και μετά την Υπουργό Νάγκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τις συστάσεις θα τις ενσωματήσω τόσο θα ήθελα πολύ να τις εσωματώσω στις συζητήσεις που θα έχουμε με τις διάφορες αρχές και φορείς όσον αφορά το θέμα του Erasmus Plus. Βεβαίως και θα πρέπει να βελτιωθεί η πράξη απαντώντας στην ερώτηση που μου έγινε φυσικά και στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα πρέπει να αξιολογήσουμε πώς υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα Erasmus Plus σε όλη την Ευρώπη για να ενσωματώσουμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα με μια σωστή ανάλυση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες για θέματα νεότητας, Φυσικά και θα πρέπει να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε την ε, καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας, να διευκολύνουμε την ε, ενσωμάτωση. Είναι το θέμα τόσο σημαντικό που πρέπει σίγουρα να ξεπεράσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και σε άλλες χώρες. Σημειώνω λοιπόν αυτήν σας την παρατήρηση και θα δω πώς μπορούμε να την ενσωματώσουμε. Κυρία Evans, ζητήσατε αν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα λάβουμε υπόψη μας και το θέμα της κατανομής αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη. Βεβαίως η παιδεία είναι εθνική αρμοδιότητα, πολλές φορές περιφερειακή, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειών, των περιοχών, με διαφορετικές παραδόσεις και όπως και στον πολιτισμό θα λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και των περιφερειών της Ευρώπης. Το Λουξεμβούργο έχει επαφές με τη Γερμανία και κυρίως με τα κρατήδια. Είναι πολύ κοντά στη χώρα μας και ξέρουμε ότι Πρόκειται για αρμοδιότητα των γερμανικών λέντερ, των κρατηδίων. Στη Γερμανία το θέμα της ε, εκπαίδευσης είναι δική τους αρμοδιότητας και συζητούμε με τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να το κρίνω εγώ. Κύριε Πρόεδρε, υπενθυμίσατε και τη μεγάλη σημασία της πολυγλωσσίας. Σήμερα, σαν Προεδρία, μπορούμε να τοποθετηθούμε εν ώψη των διαφόρων μέτρων που έχουν ληφθεί από τις χώρες. Είναι πολύ μεγάλη σημασία της πολυγλωσσίας. Μπορεί να προσφέρει στα παιδιά, στους έφηβους, στους νέους πολλά. Ξέρετε ποια είναι η θέση μου και καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας μας θα παραμείνω σταθερός στην πεποίθησή μου. Πάντα το να μαθαίνει κανείς μια παραπάνω γλώσσα είναι θετικό. Εκτός βέβαια αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες περιπτώσεις σε αποτυχία σχολική. Σε πολλά σχολικά συστήματα υπάρχουν παιδιά που μαθαίνουν δύο ή τρεις ξένες γλώσσες στο σχολείο, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και βεβαίως η μητρική τους γλώσσα είναι τελείως διαφορετική ή πολλές φορές έχουν δύο μητρικές γλώσσες. Βεβαίως σε καμία περίπτωση η εκμάθηση πολλών ξένων γλωσσών δεν θα πρέπει να αποτελέσει ε, λόγο αποτυχίας στο σχολείο. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στην ερώτηση της κυρίας Κάμερβερτ για τα πνευματικά δικαιώματα. Η Προεδρία γνωρίζει ότι η μεταρρύθμιση στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε σαν πρόκληση και όσον αφορά την κυκλοφορία και όσον αφορά την πρόσβαση των έργων σεβόμενοι τα δικαιώματα των ε, συγγραφέων, τα πνευματικά δικαιώματα και φυσικά περιμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Κυρία Τρέπελ πολιτισμός και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία μας βεβαίως και γνωρίζει ότι πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται σε πολύ πρόωρο στάδιο. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να μιλήσει για ειδικά κονδύλια βεβαίως. Από την άλλη πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια γι' αυτό και επιμένω όσον αφορά τον εγκάρσιο χαρακτήρα αυτής της πολιτικής, να στηριχτούμε στο κοινοτικό και κτημένο. και φυσικά αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί και μετά την Προεδρία του Λουξεμβούργου χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος ε, Στογεύσκη έκανε μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. ευχαριστώ. Ξέρω ότι όταν εσείς είχατε την ε, Προεδρία, ε, ήσασταν Υπουργός Πολιτισμού και οι στατιστικές ήταν πολύ σημαντικές ε, για την Προεδρία σας. Οι σχέσεις λοιπόν με την Eurostat έχουν ξεκινήσει εκ νέου έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Ξέρετε ότι το Λουξεμβούργο έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις, ε, την πρόοδο που γίνεται σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό και ξέρω ότι στις διάφορες μελέτες της Eurostat όσον αφορά την κατανάλωση, το θέμα του πολιτισμού λείπει τελείως από τις στατιστικές αυτές. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που ακούστηκε και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για τις δεσμεύσεις, για τις απαντήσεις που δώσατε και για την βούλησή σας να συνεργαστείτε στενά με την Επιτροπή μας. Είμαστε στη διάθεσή σας και φυσικά Περιμένουμε στρατηγικές πρωτοβουλίες με μεγάλη χαρά. Θα είμαστε παρόντες και στις συναντήσεις που οργανώνεται στο Λουξεμβούργο και φυσικά θα κάνω μια έκκληση για θέματα δημοσιονομικά. Ώστε να προστεθούν όχι τεράστια κονδύλια, αλλά εν πάση τουλάχιστον να μην περικοπούν. Μετά από την μεγάλη μάχη που είχαμε δώσει στο Κοινοβούλιο να έχουμε περισσότερα κονδύλια για τα θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης, να μην το ξεχνούμε αυτό. Είναι η τεράστια προτεραιότητα στο εσωτερικό των πολιτικών. Ανησυχούμε λοιπόν για την ε, περικοπή στην ε, Creative Europe και στα θέματα της αρμοδιότητάς σας που δεν είναι ακριβώς ε, δικά μας, αλλά εν πάση εκείνα που αφιερώνονται στο πλαίσιο του ορίζοντος 2020, ε, ε, σημειώνουμε περικοπές που είναι τελείως εκτός κλίμακος. Και αυτό θα εξακολουθήσουμε να το, το συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μετά την αποχώρησή σας. Ε, επομένως υπολογίζουμε στην συνεχιζόμενη υποστήριξή σας και στη συνεργασία σας ε, ευχαριστούμε, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία για την Προεδρία. Colleghi, non fuggite, don't go out because... Μην διαφεύγετε, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. And so, we continue with the ε, ε, Συνεχίζουμε λοιπόν με την ε, γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού. Θα παρακαλούσα καταρχάς να συναδέλφους να παραμείνουν στην αίθουσα, γιατί αυτό το τελευταίο θέμα είναι σημαντικό. Πρόκειται για το σχέδιο γνωμοδότησης επί των θεμάτων προϋπολογισμού του κυρίου Σδρογεύσκη και για τους, ε, τις τροπολογίες. Ο κύριος Σιασδρογεύσκη θέλει κάτι να πει παρότι έχουμε μείνει λίγοι αλλά καλοί όπως λένε. Θα είμαι πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Θα σας ε, ενημερώσω για το τι θα συμπεριληφθεί στην γνωμοδότηση. Πολύ καλά φαίνονται τα πράγματα για το 2016. Βλέπω αύξηση των πληρωμών, μείωση τη ανάληψη υποχρεώσεων. Αυτό αφορά το Erasmus, 30%, το Creative Europe, αύξηση και εκεί. Και ελπίζω να υπάρχει και μία παρόμοια αύξηση σχετικά με τις πληρωμές για τα υπόλοιπα προγράμματα. Επίσης υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές του προηγούμενου έτους. Οι αυξήσεις είναι λιγότερες και μάλιστα ένα πρόγραμμα υπέστη και μείωση κατά 2% στα πλαίσια του Creative ε, Europe. Αυτό που μας ανησυχεί σχετικά με το 2016 είναι ότι δεν υπάρχει αποθεματικό για τα πιλωτικά προγράμματα πιστεύω πως πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερο αποθεματικό και περισσότερες δυνατότητες για την προσθήκη και άλλων πιλωτικών προγραμμάτων πέραν των φυσταμένων. Πέντε σημαντικά σημεία εγκρίθηκαν τον Ιούνιο. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το Erasmus Plus, όμως όπως τόνισε και η συνάδελφος λίγο νωρίτερα, χρειάζεται να ε, πολεμήσουμε έτσι ώστε να ε, γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή του προγράμματος, να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη ευελιξία. Σχετικά με τα πολυμέσα 010505, να τονίσω ότι το Euronet Plus είδε μείωση στις ε, καθυστερήσεις πληρωμών, αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Τέλος, προτείνουμε να μην μειωθούν οι οικονομικοί πόροι για τα προγράμματα των ε, πολιτών. και να προστατευτούν. Οι πόροι η διαθέσιμη πόρη για το 2016. Όπως είπα, είμαστε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι με την γενικότερη αύξηση που έχει παρατηρηθεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε τον κύριο Ζρογεύσκη για την ε, έκθεση αυτών των στοιχείων. Ε, Μόργανο παρακαλώ να πω σύντομα ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις αυτές. Πρέπει να επιμείνουμε σε κάποια θέματα διότι το να διακινδυνεύσουμε, στο να περιοριστούμε στα τρέχοντα, δεδομένης της κατάστασης, είναι ανεπαρκές. Έχουμε, πιστεύω, τη δυνατότητα μαζί με την Επιτροπή να καθορίσουμε κάποιες προτεραιότητες για να αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον ευρωσκεπτικισμό σε κάποια στοιχεία φονταμενταλισμού διαφόρων ειδών που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη και μέσω της, ε, των δεσμεύσεων του προεμπολογισμού ε, νομίζω ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις προθέσεις μας αυτές σε απτές δράσεις, σε πράξεις. Η Έλγα, παρακαλώ. Να πω ότι δεν δέχομαι την μείωση αυτών των γραμμών του προπολογισμού, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την Europe for Citizens. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν έχει κανένα νόημα να περικοπούν αυτά τα κονδύλια, ιδιαίτερα όταν ε, λέμε ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε τους ε, πολίτες και να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες δέσμευσης. Πραγματικά εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε περαιτέρω περικοπών. Είναι κόκκινη γραμμή για μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε περαιτέρω περικοπές. Είναι αντιπαραγωγικό αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Προφανώς υπό το φως των όσων συνέβησαν στο Συμβούλιο και συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή και των σκιωδών πρέπει να ζητήσουμε σημαντικές αυξήσεις για να δηλώσουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε προς τα πίσω αλλά πρέπει να πάμε προς τα εμπρός. Και συμφωνώ και για την red line, λέει η πρόεδρος. Για παράδειγμα βλέπω ότι περικόπτεται στο Creative Europe το οριζόντιο της νέας facilities του νέου μηχανισμού που θα ξεκινήσει από το 2016. Ήδη ξεκινάει λοιπόν με μείωση. Πρέπει λοιπόν να επιτηρήσουμε ότι δεν θα συμβούν αυτά. Όπως και για το Europe Citizens. Νομίζω ότι μαζί με την Επιτροπή Προεπολογισμού λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά αυτά τα θέματα και σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στην Επιτροπή Πολιτισμού αυτό θα είναι 15 Σεπτεμβρίου και προθεσμία 25 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι για την υποβολή τροπολογιών. Με αυτό θεωρώ ότι μπορώ να κλείσω την πρωινή συνεδρίαση. Θα τα πούμε στις 3 η ώρα με τους δύο επιτρόπους και θα παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους και τους συντονιστές των ομάδων διότι δώσαμε μάχη για να έχουμε αυτές τις συναντήσεις στρατηγικής πλέον σημασίας να είναι όλοι παρόντες θα τα πούμε τρεις η ώρα. Ευχαριστώ.